είναι περισσότερο που αυτά τα νούμερα ε, δεν περιλαμβάνουν καν ε, τον, τον πόνο και τη θλίψη των ανθρώπων που χάνουν τους δικούς τους. Ευχαριστώ. Ολοκληρώνω τις συζητήσεις για την ε, πλημμύρα. Να σας ενημερώσω ότι από την ομάδα έλαβα τον κατάλογο ορισμών βουλευτών που ορίζονται σε κοινοβουλευτικές ομάδες. Θα υπάρχουν στα πρακτικά και αν δεν υπάρξουν αντιρρήσεις οι τοποθετήσεις αυτές θα εγκριθούν. Επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη. Έκθεση ποδηματά για την υλοποίηση ενισχυμένη